Έχουμε την ημερήσια διάταξη. Βάσει του κανόνα 142 και σε σχέση με την δημοκρατία της Βενεζουέλας και την αλληλεία στα ύδατα της Γαλλικής Γκουγιάνας έλαβα ένα αίτημα για κατεπήγονσα διαδικασία σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου και μια ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης. Πρόκειται για την κατεπήγουσα ε, διαδικασία σχετικά με την αλληλεία στα ύδατα της Γαλλικής Γουγιάνας από τους πράσινους ε, Ευρωπαία, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη